Bien, mesdames, messieurs, chers collègues. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, με συγχωρείτε για την άλλη φορά καθυστέρηση, αλλά τα ρολόγια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δυστυχώς ε, κάθε εβδομάδα φαίνεται να καταγράφουν μεγαλύτερη καθυστέρηση, κάτι που δεν ε, είναι καλό σημάδι και πρέπει, ξέρετε, να μην επιδεικνύουμε ότι καθυστερεί η Ευρώπη και αυτό θα έχει πολύ άσχημο αντίκτυπο ε, στις εργασίες μας και ιδίως στις εξωτερικές υποθέσεις. Λοιπόν, ας ε, ξεκινήσουμε με την ε, συζήτηση της ε, έκθεσης ε, του κυρίου Γκουαλτιέρη που έχει να κάνει με την ε, κοινή πολιτική ασφαλής και άμυνας μετά την άνοιξη ισχύω της συνθήκης της Λισαβόνας. Πρόκειται για γενική έκθεση, έναν απολογισμό της και της και ΕΠΑ, γιατί θέλουμε να δούμε πώς τεθήκαν σε εφαρμογή τα κεκτημένα της συνθήκης της Λισαβόνας και πώς μετά από ένα έτος της θα σε ισχύ τη συνθήκη ετέθηκαν σε εφαρμογή οι νέε διατάξει. Έτσι λοιπόν, θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκουαλτιέρη, ο οποίο ε, θα μα ε, παρουσιάσει την έκθεση αυτή και κατόπιν θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Ο κύριο ε, Γκουαλτιέρη συμμετέχει και στην Επιτροπή ΑΦΚΟ και θα πρέπει να μας εγκαταλείψει στις 10.30. Έτσι λοιπόν έχουμε λιγότερο από μία ώρα για το ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα σας αναφέρω τα κυρία σημεία της έκθεσης ε, που θα παρουσιάσω την επόμενη Δευτέρα. Θα λάβουν λοιπόν το κείμενο οι συνάδελφοι σε λίγες μέρες, αλλά ήθελα να έχουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων πριν παρουσιάσω ένα σχέδιο κειμένου, έτσι ώστε να μπορέσω να ακούσω διάφορες προτάσεις ε, και ενδείξεις και να έχουμε μια πρώτη τελεγή αποψίων επί κάποιων σημείων που θα συμπεριληφθούν στην εκθεσή μου. Το μέγεθος ε, της ε, έκθεση το υπενθύμησε ο κ. Ντενσεν. Εγώ ήθελα και το θέμα της εκθεσής το ο κ. Εγώ ήθελα να κάνω μια εκθέση που θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όμως δεν θα ήθελα να λέω τα πάντα επί παντός επιστητού. Έτσι λοιπόν θα σας παρουσιάσω τώρα ένα δύο ε, δείκτη και σε αυτόν θα σας παρουσιάσω κάποια σημεία που θεώρησα ότι είναι πιο προβληματικά ή που χρειάζεται να σκεφτούμε περισσότερο και που τοποθετούνται ε, στο ευρύτερο φάσμα μεταξύ των ε, θεμάτων που έχουμε σήμερα επιτάπητος, της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης, των δομών και των ε, ικανοτήτων ε, τη ΚΕΠΑ και από την άλλη της καινοτομίας της συνθήκης της Λισαβόνας ε, και του διεθνού περιβάλλοντος που είναι ανεξελίξη. Η έκθεση διαρθρώνεται σε έξι κεφάλαια που έχουν όλα στο επίκεντρο τη σχέση μεταξύ της ΚΕΠΑ ή της διάστασης της ασφάλειας και των διάφορων πτυχών της εξωτερικής δράσης της Ένωσης. Αυτό είναι ε, το κύριο νήμα που ακολουθεί η έκθεση και η συνολική προσέγγιση είναι μία απέτηση που γεννάται από τις εξελίξεις στο διεθνές πλαίσιο, δηλαδή από τις νέες διαστάσεις της ασφάλειας ε, που παρουσιάζονται σε διεθνές επίπεδο είτε είναι ένα στοιχείο που εγώ πιστεύω ότι είναι στο επίκεντρο των καινοτομιών, των ε, πλέον αλλά και λιγότερο προφανών της συνθήκη τη Λισαβόνα. Τα κεφάλαια είναι και πάει η ασφάλεια και εξωτερική δράση, ασφάλεια και άμυνα, εξωτερική ασφάλεια και εσωτερική ασφάλεια, ασφάλεια μέσω των επιχειρήσεων, ασφάλεια εσωτερική σχέση, ασφάλεια και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα, για να σας παρουσιάσω ποια είναι τα κυρία σημεία. Σε ό,τι αφορά στο πρώτο, που είναι η ανάλυση της σχέσης της ΚΕΠΑ και των άλλων διαστάσεων της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Άνωσης, ε, δηλαδή ε, της ε, πολιτικής άμυνας και ασφάλειας, αλλά όχι μόνο της κοινή πολιτικής άμυνας και ασφάλειας. Έχουμε εδώ την καινοτομία της Συνδίκης της Λισαβόνας. Ε, και είναι ε, το οι πιο βαθιές καινοτομίε πιο προφανείς, που έχουν να κάνουν με την ε, ΕΠΑ και την ΚΕΠΑ. η ΚΕΠΑ είναι, ε, συγγνώμη, ΕΠΑ είναι τμήμα της ε, ΚΕΠΑ και όπως ε, κεπα υπήρχε στη συνθήκη και αποκεφαλίστηκε κατά κάποιο τρόπο από συγκεκριμένου ε, στόχους όπως είχαμε στην παλιά συνθήκη. Εδώ με το 2011 που είχαμε τους συγκεκριμένους στόχους της, εξωτερικής, της κοινής εξωτερικής πολιτικής ασφαλής και άμυνας. Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας. Εδώ ε, το βάζουμε αυτό το θέμα στο κεφάλαιο 22 και εκεί αναφερόμαστε σε όλους τους στόχους της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιε είναι οι συνέπειες ε, αυτού του στοιχείου, όπω και άλλων στοιχείων, δηλαδή αναδιατύπωση του άρθρου 40, του άρθρου 40, γιατί το παλιό άρθρο 47 ανέφερε ποιο είναι το όριο μεταξύ των αρμοδιοτήτων της ΚΕΠΑ και των κοινοτικών αρμοδιοτήτων. Και στη συνέχεια το δικαστήριο είχε θέσει τις ε, νομικές βάσεις των συγκεκριμένων δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επίσης ε, είχαμε και την ανάλυση ε, και πιο πρόσφατων αποφάσεων, όπως για τα ελαφρά όπλα. Όλα αυτά μας οδηγούν ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την ασφάλεια έναν οριζόντιο στόχο της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, ε, περισσότερο από ότι ένα στόχο της συγκεκριμένης πολιτικής. Έτσι, λοιπόν, ε, η ΚΕΠΑ και η ΕΠΑ, πέρα από ξεχωριστές πολιτικές, είναι περισσότερο εργαλεία ε, συνολική δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φυσικά αυτό θέτει προβλήματα, νομικά προβλήματα, δηλαδή προβλήματα για τη νομική βάση γιατί έχουμε διαφορετικέ νομικέ βάσει στο εσωτερικό όμω πολιτικών που τελικά πρέπει να δράσουν από κοινού. Και έχουμε και οργανωτικά και πολιτικά προβλήματα. Έτσι λοιπόν, αυτά αναφέρονται στο κεφάλαιο που έχει να κάνει με ε, τη ε, συσχέτιση ε, της ΚΕΠΑ και των υπόλοιπων ε, ε, στοιχείων της εξωτερικής δράσης και εκεί αναφερόμαστε σε μία διαχείριση που θα βασίζεται στις σχέσεις της ΚΕΠΑ που πρέπει να έχει μία ιεραρχική σχέση με την υπατή εκπρόσωπο είτε με τις άλλες υπηρεσίες εξωτερικής δράσης, με τις περιφερειακές δηλαδή υπηρεσίες είτε με τις δομές της ε, πολυμερής Και ο στόχος ε, είναι να καταλήξουμε στην διαχείριση κρίσεων, αλλά βάσει ε, μιας συσχέτισης αυτών των στοιχείων. Κατόπιν έχουμε το πρόβλημα της ενίσχυσης ε, των δυνατοτήτων του επιχειρησιακού σχεδιασμού της πολιτικής αυτής. Κατόπιν έχουμε την ε, μεταφορά στην εξωτερική υπηρεσία ε, των ε, υπηρεσιών διαχείρισης της, του μηχανισμού σταθερότητας. Έχει γίνει μια συζήτηση μεταξύ Κοινοβουλίου και της, της κυρίας Άστον και της Επιτροπής. Έτσι λοιπόν υποστηρίζουμε το να υπάρχει μια διοργανική δομή όπου θα βρίσκουμε από κοινού τα στοιχεία της διαχείρισης των μη στρατιωτικών επιχειρήσεων μαζί με τις δομές της Επιτροπής της Εξωτερικής Υπηρεσίας. Και έτσι θα γίνεται μια καλύτερη διαχείριση των μη στρατιωτικών επιχειρήσεων. Αυτά είναι σημαντικά στοιχεία αυτού του κεφαλαίου. Και επίσης εξετάζουμε το πώς θα υπάρξει ολοκλήρωση μεταξύ διαφορετικών δομών και εργαλείων, όχι μόνο στρατιωτικών και μη στρατιωτικών στο εσωτερικό της ΚΕΠΑ, αλλά ε, και στρατιωτικών και μη στρατιωτικών στοιχείων της ΚΕΠΑ και άλλων ε, φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διαχείριση των κρίσεων. Υπογραμμίζουμε το παράδειγμα του Πακιστάν, ε, όπου είδαμε ότι υπήρχε πολύ μεγάλη διαφορά στη διαχείριση σε σχέση με την περίπτωση της IT's. Δηλαδή είχαμε ε, συνεισφορές από μεμονωμένα κράτη στην IT ενώ στην περίπτωση του Πακιστάν υπήρξε ένα συντονισμός για τη χρήση των στρατιωτικών μέσων στο πλαίσιο μια δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στην περίπτωση αυτή δεν ήταν ε, μια αποστολή, ε, αλλά ε, ήταν μια καθαρά μη στρατιωτική, δεν ήταν αποστολή άμυνας και ασφαλής, ήταν καθαρά μη στρατιωτική αποστολή, αλλά χρησιμοποίησαμε και στρατιωτικά μέσα. Το δεύτερο κεφάλαιο, θα είμαι πιο σύντομο τώρα, αφορά τη σχέση μεταξύ ασφάλειας και άμυνας. Εδώ από πολιτική σκοπιά υπογραμμίζουμε ότι η έμφαση στη συνολική προσέγγιση, στην αγκαιότητα να έχουμε διαφορετικά μέσα στρατιωτικά και μη στρατιωτικά και πολιτικά, δεν πρέπει να σημαίνει ότι η Ευρώπη εγκαταλείπει τη δυνατότητα να έχει κλασικά μέσα χρήση στην περίπτωση της άμυνας. Έτσι λοιπόν τονίζουμε πόσο σημαντικό είναι να έχουμε και στρατιωτικά μέσα στα πλαίσια αυτής της συνολικής προσέγγισης. Εδώ έχουμε κάποιες συγκεκριμένες πτυχές που αναφέρονται. Τονίζουμε την απέτηση μιας ε, ενεργούς εκπόνησης της ε, ρήτρας αμοιβαίας ε, αρρωγής και Έχουμε και το ζήτημα, το Operational Headquarters, ε, τη δυνατότητα να ενισχύσουμε το κέντρο επιχειρήσεων που έχουμε σήμερα, είτε με διάμεσα στάδια, είτε μέσω της προοπτικής να έχουμε ένα πραγματικό τέτοιο επιχειρησιακό κέντρο και εκεί να έχουμε και μία πτυχή μη στρατιωτική με σημαντικές διαστάσεις. Ανοίγουμε δηλαδή ένα προβληματισμό και για το κόστος ε, και η απάντηση της κυρίας ε, Άστον δεν εκφράζει αντίρρηση επί της αρχής. Ε, αυτό είναι θετικό, αλλά υπογραμμίζει το ότι πρέπει να γίνει μια ανάλυση κόστους ωφέλους, θέτοντας και το πρόβλημα του κινδύνου με απρόσθετη δομή στις πέντε εθνικές δομές να είναι μια αποτελεσματική. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ληφθεί μια πολιτική απόφαση προς αυτή την κατεύθυνση. Κατόπιν ε, έχουμε το θέμα για τον ε, οργανισμό άμυνας υπάρχει και ένα τμήμα που αφορά την απέτηση να ενισχύσουμε ε, την εσωτερική αγορά άμυνας ως προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την αναδιάρθρωση της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας Άμυνας. Έχουμε και ένα τμήμα για τα battle groups Εκεί υπογραμμίζονται τα προβλήματα της χρήσης τους, υπερασπίζουμε αυτό το μέσο, αλλά αναλύονται δυνατότητες να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τα battle groups, είτε ε, μέσω μεταρρύθμισης του μηχανισμού των Αθηνών, που επιτρέπει να χρησιμοποιείται ένα τμήμα των δαπανών μέσω του κοινού κόστους, είτε μέσω μιας διαφοροποίησης των battle groups και του ε, καθορισμού ενός battle group που να αναλαμβάνει πιο διαφοροποιημένα καθήκοντα σε σχέση με τα πιο συγκεκριμένα καθήκοντα που έχει σήμερα για της ε, ταχείας επέμβασης σε έντονες σειράξεις και με δυνατότητες ε, που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το battle group και σε διαφορετικές συνθήκες. σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο για τη σχέση εξωτερικής και εσωτερικής ασφάλειας. Τονίζουμε το πόσο λιλένδετες ε, είναι οι δύο διαστάσεις αυτές. Αναφέρουμε και την ρήτρα αλληλεγγύης της συνθήκης, ότι καλύπτουμε και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας με τις αποστολές. Αναφέρουμε το πρόβλημα ε, στο ότι έχουμε δύο διαφορετικά νομικά πλαίσια, το κοινοτικό αλλά και το υποκείμενο στην ΚΕΠΑ και φυσικά είναι απέτηση να ε, ε, διατηρήσουμε ως και την κοινοτική μέθοδο. Ε, αναφέρουμε την ε, δυνατότητα να ανισχύσουμε το διάλογο μεταξύ ΚΟΖΙ και ΚΟΠΣ προκειμένου να μπορέσουμε να χρησιμοποιούμε διαφορετικά μέσα όταν υπάρχουν ε, προκλήσεις στην ασφάλεια, γιατί πολλές φορές είναι δύσκολο να τις κατηγοροποιήσουμε σε εξωτερικές και εσωτερικές απειλές. Κατόπιν, ε, δεν κάνω μια ανάλυση όλων των αποστολών, αλλά αναφέρω κάποιους προβληματικούς κόμβους και κάποια πιο γενικά προβλήματα. Παραδείγματο χάρη για τη χρηματοδότηση, τονίζω την ε, αναγκαιότητα να έχουμε το ε, ταμείο Startup ε, και αναφέρομαι και στο Μηχανισμό των Αθηνών και αναλύω τις αποστολές όπου αναφέρεται, ε, εμφανίζεται με πιο προβληματικό τρόπο η σύνδεση μεταξύ στρατιωτικής και πολιτικής στρατηγικής. Νομίζω ότι αυτό το τμήμα δεν είναι δυνατό να αναπτυχθεί όπως πρέπει, όπως δεν αναπτύσσω και το τμήμα για τις εταιρικές σχέσεις και το τελευταίο κεφάλαιο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την ασφάλεια. Εκεί αναλύω τις καινοτομίες συνθήκης της Λισαβόνας ε, και τις καινοτομίες που προέκυψαν από τη Συμφωνία της Μαδρίτης και από τη δήλωση της ε, εκπροσώπου και τα προβλήματα που έχουν ε, προκληθεί κατόπιν της ολοκλήρωσης της δυτικής συνδιάσκεψης και αναφέρομαι σε προβλήματα που είναι γνωστά σε όλους. Δεν χρειάζεται λοιπόν να τα αναφέρω τώρα. Έτσι λοιπόν η δομή της έκθεσης είναι αυτή που σας ανέφερα. Θέλω πάρα πολύ να λάβω τα δικά σας σχόλια και ενδείξεις. Με ενδιαφέρουν τα μάλλα. Ευχαριστώ. Bien, merci beaucoup. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν πολλοί που θέλουν να πάρουν το λόγο. Κύριος Καλέρα και το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ πολύ ε, αγαπητέ συνάδελφε κύριε Γκουαλτιέρη για όλα αυτά που μας είπατε. Νομίζω ότι με την ε, δομή που παρουσιάσετε θα έχουμε τελικά μια πολύ καλή έκθεση. Ε, επί της ουσίας και σε επίπεδο αρχής συμφωνώ με τη δομή, τα διάφορα κεφάλαια, τα μεμονωμένα θέματα που είναι πράγματι περίπλοκα. Μετά τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας, ε, θυμάμαι ότι είχαμε ε, υψηπετείς ε, φιλοδοξίες ε, και πριν από τη Λισαβόνα. Και αυτό που τελικά προέκυψε από τότε πριν από τη συνθήκη και αυτό που προέκυψε μετά τη συνθήκη υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Θυμάμαι τι αποφασίστηκε σε ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τότε ε, όπου αποφασίστηκε για πολλές ε, και μεγάλες και μικρές αποστολές ή ε, το δυναμικό που θα προέκυπτε. Προφανώς υστερούμε όσον αφορά αυτές ε, τις αποφάσεις και νομίζω ότι η νέα συνθήκη μας δίνει τη δυνατότητα σε επίπεδο πολιτικής βούλησης να μειώσουμε λιγάκι το χάσμα ανάμεσα σε φιλοδοξίες και πραγματικότητα. Τα θέματα που θίξατε ενδείκνυνται για να επιτύχουμε το στόχο μας. Πρόκειται λοιπόν για την ενίσχυση των ε, δυνατοτήτων και του δυναμικού Πρόκειται για το ότι οφείλουμε να ορίσουμε πού θα υπάρχουν αυτές οι μόνιμες δομές συνεργασίας, Permanent Structure Corporations, και επίσης πρόσφατα λάβαμε και πιο συγκεκριμένες προτάσεις. Υπάρχει μια γαλλο-σουηδική επιστολή για pooling and sharing ε, το οποίο βασικά εγκρίθηκε από το Συμβούλιο το Δεκέμβρη και αυτή τη στιγμή υπάρχει και άλλο ένα έγγραφο του τριγώνου της Βαϊμάρης, το οποίο και αυτό συζητιέται. Και νομίζω εκεί γίνονται περισσότερες σκέψεις, συνέχεια των σκέψεων του τι μπορεί να ε, βελτιωθεί στην πράξη. Ε, στηρίζω αυτό που είπατε για, το, για τα την επιχειρησιακή έδρα, headquarters, και εγώ πιστεύω ότι χρειαζόμαστε το μηχανισμό της Αθήνας και σε σχέση με αυτό αναφέρατε το θέμα του κόστους γιατί νομίζω όσοι λειτουργούν τα πράγματα αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να παραταθούν στο δίνεκες Είναι λοιπόν αλήθεια ότι πρέπει να δούμε λιγάκι πώς ε, ακριβώς ε, θα λειτουργήσει η ενιαία αγορά για τα ε, αμυντικά εμπορεύματα, για τα αμυντικά αγαθά. Ε, πράγματι ε, πρέπει τώρα να ασχοληθούμε το θέμα αυτό γιατί εκείνο που ενδιαφέρει είναι να μην δαπανάμε περισσότερα χρήματα από όσα πρέπει. Και εάν υπάρξει τελικά ενιαία αγορά, προφανώς θα πρέπει να πέσει η τιμή των προϊόντων και να υπάρχει και καλύτερη χρήση. Τούτο αναμφίβολα θα έχει θετική επίδραση στο κόστος. Αναφερθήκατε σε μια συνολική προσέγγιση, τη συνεργασία του αστικού και του στρατιωτικού σκέλους. Αυτό ε, παραμένει ένα από τα θεσμικά πλεονεκτήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τον ΝΑΤΟ. Θεωρώ λοιπόν ότι όσον αφορά αυτό το σημείο επαφής ανάμεσα στην εξωτερική και την εσωτερική ασφάλεια, Εκεί, σε αυτό το θέμα, πρέπει να δούμε ε, πώς θα να υπάρχει καλύτερη λειτουργία. Δηλαδή, οι αρμόδιοι φορείς ε, να μπορούν να επιτύχουν τη βέλτιστη δυνατή συνεργασία. Μέχρι τώρα υπήρχε σαφής διαχωρισμός σε εθνικό επίπεδο, διότι οι απειλές που αντιμετωπίζουμε κυρίως από τον τομέα της ε, τρομοκρατίας, αυτές οι απειλές δεν κάνουν το διαχωρισμό της εσωτερικής και της εξωτερικής ασφάλειας. Μπορεί ιστορικά να ανάγονται στο επίπεδο της ε, εξωτερικής ασφάλειας, αλλά αν δει κανεί ε, την έκταση των απειλών αυτών, καταλήγει στο ότι θα μπορούσε μάλιστα να μιλήσει και για κατάσταση πολέμου. Είναι λοιπόν σημαντικό να υπάρχει σαφής διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων και ε, κάποια μορφή συνεργασία. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα όμω που δεν το θίξατε και νομίζω ότι πρέπει να συμπεριληφθεί. Πρόκειται για τη θέση ανάμεσα στην πολιτική ασφάλεια και την αναπτυξιακή πολιτική. Αυτό είναι ένα θέμα που συζητιέται όλο και περισσότερο λόγω του ότι σε πολλέ χώρε του τρίτου κόσμου εμφανίζονται κρίσει. Βλέπουμε και τι συμβαίνει και στη Βόρεια Αφρική. Έτσι λοιπόν εδώ τίθενται τόσο θέματα ασφάλειας όσο και ανάπτυξης. Και γι' αυτό το λόγο οφείλουμε να μεριμνήσουμε να είναι συνεπείς οι πολιτικές μας. Δηλαδή να μην προβαίνουμε σε ένα διαχωρισμό όπου η αναπτυξιακή πολιτική να είναι για τους ε, καλούς πολίτες και η πολιτική ασφάλειας για τους άλλους που έχουν ε, άλλες προθέσεις. Όχι, δεν είναι σωστό αυτό. Εγώ νομίζω ότι όταν χαράσουμε μια πολιτική απέναντι σε μια χώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να χαράσει την ίδια πολιτική, ε, είτε κάτω από το μανδύα της πολιτικής ασφάλειας, πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτική ανάπτυξης, γιατί σε τελική ανάλυση οι πολίτες αυτών των ε, χωρών θεωρούν ότι είναι πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης άσχετα από το Μανδύα. Ως εκ τούτου πρέπει να δίνουμε μια σφαιρική εικόνα της πολιτικής μας. Χαίρομαι λοιπόν που μας ε, καταθέσατε αυτό το πρώτο σχέδιο. Η δομή είναι καλή και πάνω σε αυτή τη βάση μπορούμε να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε ο κύριος Πασκού. Well, Σας ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω και εγώ ότι η προσέγγιση είναι καλή και είναι θετικό ότι προτού ξεκινήσετε τη σύνταξη της έκθεσης αυτής, σε στρατηγικό επίπεδο ήρθατε σε επαφή μαζί μας προκειμένου να καταφέρουμε να κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων και να καταλήξουμε σε κάποιες κοινέ ιδέες βάσει των οποίων πιστεύω ότι μπορείτε να χτίσετε την έκθεσή σας. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό αποτελεί ένα πολύ καλό προηγούμενο. Να πω επίσης ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε μια κάποια ισορροπία ανάμεσα στο θεσμικό, ρυθμιστικό πλαίσιο, πραγματικότητα, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένας οργανισμός, όπως ξέρετε, ιδιαίτερα πολύπλοκος, με πληθώρα κανόνων, και ανάμεσα στην πραγματικότητα που βλέπουμε επιτόπου, Και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω την πρώτη, φράση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την ασφάλεια «Η Ευρώπη ουδέποτε υπήρξε τόσο ευήμερη, τόσο σταθερή, τόσο ασφαλής, ε, ποτέ στην ιστορία της». Με όλα αυτά τα οποία πρόκειται να συμβούν ή συμβαίνουν στη Βόρεια Αφρική, μπορούμε να πούμε επομένω ότι η φράση αυτή ακόμα ισχύει και ότι θα ισχύει και στο μέλλον. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να κρατήσουμε μια κάποια ισορροπία ανάμεσα σε όλα αυτά τα οποία ισχύουν από θεσμική πλευράς και ανάμεσα στην πραγματικότητα από την άλλη. Την πραγματικότητα πολλές φορές μας εκπλήσει. Ανάμεσα στην άμεση αυτή εξέλιξη των πραγμάτων. Και πολλές φορές βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφορες εξεγέρσεις, τις οποίες δεν μπορούμε καν να προβλέψουμε, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να αντιδράσει σε σχέση με αυτές. Κανείς δεν μπορεί να αντιμετωπίσει με μονομένα τις κρίσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Βόρεια Αφρική. Αντίθετα, θα πρέπει να έχουμε μία κοινή προσέγγιση στην πρόκληση αυτή. Η στάση μας δηλαδή να μην είναι κατακαιρματισμένη. Όταν επανέλθουμε μετά στο ζήτημα το ρυθμιστικό, το θεσμικό, όταν θα πρέπει να ασχοληθούμε δηλαδή με αυτό το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο σαφώ πρέπει να αντιμετωπίσουμε, θα πρέπει τότε να καταφέρουμε να πετύχουμε την μέγιστη δυνατή ευελιξία, προκειμένου να μπορούμε εμεί με ευελιξία να ανταποκρινόμαστε στι μεγάλε προκλήσει. Πρώτον αυτόν. Δεύτερον, θα πρέπει να καταφέρουμε να προωθήσουμε μία κάποια κοινή προσέγγιση περιφερειακή όσον αφορά τις κρίσεις αυτές και έπειτα να πόκειται στις χώρες να αποφασίσουν αν θα εμπλακούν ή όχι σε μονομένες επιχειρήσεις. Δεν θα πρέπει όταν αποφασίσουμε για το θεσμικό πλαίσιο να ξεχνάμε το ότι ουσιαστικά αυτό το οποίο θέλουμε να πετύχουμε είναι την ε, μέγιστη δυνατή αποτελεσματική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή την ισορροπία λοιπόν θα πρέπει να πετύχουμε σε όλες τις πτυχές της έκθεσής σας και χαίρομαι πάρα πολύ που προτού συντάξετε την έκθεσή σας ήρθατε πρώτα σε επαφή με εμά. Θεωρώ ότι ήταν μια πολύ καλή στρατηγική προσέγγιση. Σας ευχαριστούμε ο κύριος Βανόρντεν. Um, um Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως γνωρίζετε, εγώ έχω ένα διαφορετικό σημείο κίνησης, οι περισσότεροι ε, από τους περισσότερους συναδελφούς μας. Από ό,τι φαίνεται εσείς, βλέπετε ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι ένας φυσιολογικός στόχος, επομένως τα πάντα αποτελούν ένα βήμα παραπάνω προς την κατεύθυνση αυτή. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό το στόχο της πολιτικής ολοκλήρωσης. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κάνει χρήσιμα πράγματα, επικεντρωνόμενη όμω σε άλλες πολιτικές, όπως τον οικονομικό τομέα. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν χωρίζουν οι δρόμοι μας ήδη από την αρχή ως προς αυτό. Και το πρόβλημα είναι ότι εσείς κάθε φορά ψάχνετε μία κάποια δικαιολογία, μία αιτιολόγηση για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσπαθείτε παντού να βρείτε ένα ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από ό,τι φαίνεται πρόκληση για σας είναι να καταφέρετε κάθε φορά να δείτε πού βρίσκεται η προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βέβαια μιλάμε για πραγματική προστιθέμενη αξία και όχι για θεωρητική προστιθέμενη αξία ή για εφάνταστη προστιθέμενη αξία. Και από ό,τι φαίνεται πάρα πολλές φορές ε, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει κάπως τον εαυτό της και στις χώρες της την προσέγγιση αυτή της ολοκλήρωσης, τη συνεκτική αυτή προσέγγιση στα πράγματα. Δεν νομίζω όμως ότι ισχύει κάτι τέτοιο στην πραγματικότητα και ούτε πρόκειται να αλλάξει η προσέγγιση μας, η προσέγγιση των κρατών μελών σε σχέση με διάφορες προκλήσεις που θα έχουμε στο μέλλον. Θεωρώ ότι η προσέγγιση αυτή της ολοκλήρωσης δεν είναι κοινή για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δημιουργούμε πάντως παρόλα αυτά το μύθο αυτό ότι κάτι ιδιαίτερο συμβαίνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι η συμβολή της μπορεί να αποτελέσει κάτι ξεχωριστό. Και θα πρέπει βέβαια να παραδεχθούμε ότι πολλές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρονται περισσότερο για την ε, διατήρηση του ΝΑΤΟ ως ε, αποτελεσματική στρατηγική ε, απάντηση στα προβλήματα ασφάλειας και ενδυναμώνουν ουσιαστικά κάτι τέτοιο με διμερείς συμφωνίες. Επομένως, το Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, έχει πλέον διμερείς συμφωνίες με τη Γαλλία, αν μπορείτε να το φανταστείτε, και χαίρομαι πάρα πολύ που ισχύει κάτι τέτοιο αλλά εξίσου ενδιαφέρον ότι και η Γερμανία θέλει να συνάψει μία διμερή συνθήκη με το Ηνωμένο Βασίλειο. Επομένω, έχω την εντύπωση ότι έχουμε το ΝΑΤΟ, το οποίο αποδυναμώνει και περιθεροποιεί ουσιαστικά την δική μας την συμβολή και επιπλέον έχουμε και διάφορες διμερείς διευθετήσεις και συμφωνίες. Επομένως δεν είμαι πεπισμένος, δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς πού μπορεί να δραστηριοποιηθεί τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα σε όλη αυτή τη δομή. Θεωρώ ότι πρόκειται για μια απλή πολιτική βούληση αστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέλοντας να πετύχει τον απότερο στόχο της πολιτικής ολοκλήρωσης και θέλοντας να μπορεί να δραστηριοποιείται και ίδια με πυγμή στο διεθνές προσκήνιο. Μου προκαλεί ανησυχία όταν λέτε ότι θα πρέπει να εργαστούμε από κοινού για την ρήτρα της αμοιβαία υποστήριξης, ενίσχυσης. Γιατί ξέρετε ότι στα πλαίσια της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας λέμε ότι θέλουμε να αποφύγουμε τις επικαλύψεις. Βέβαια, ο σημαντικότερος οργανισμός για την ε, αμοιβαία υποστήριξη όταν πραγματικά προκύπτει ανάγκη είναι βέβαια το ΝΑΤΟ. Και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς πιστεύω ότι θα καταφέρει να συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτό χωρίς να στείλουμε παράλληλα κάποια σήματα τα οποία θα προκαλέσουν σύγχυση, ενώ θα πρέπει ουσιαστικά η στάση μας να είναι ξεκάθαρη. Αναφερθήκατε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα όντω μπορεί να είναι χρήσιμο σε κάποιου τομεί, πάντω δεν είμαι πεπισμένο για την ενδυνάμωση τη εσωτερική αγορά στην άμυνα και ότι αυτό αποτελεί προπόθεση για την αναδιάρθρωση τη ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Και πάλι εδώ πέρα βλέπω ότι θέτουμε έναν απότερο θεωρητικό στόχο για να καταλήξουμε μια μέρα σε μια ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει μάλλον να προστατεύσουμε τις δικές μας εθνικές αμυντικές βιομηχανίες πρώτα, αυτές που είναι στρατηγικής και ζωτικής σημασίας, αυτές οι οποίες είναι πολύ σημαντικές από οικονομικής πλευράς για τις δικές μας τις χώρες. Και αυτό που βλέπουμε πολύ συχνά είναι ότι οι διασυνδέσει πρέπει να πετύχουν μεταξύ του οι αμυντικέ βιομηχανίε δεν είναι μεταξύ των κρατών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών και τρίτων χωρών. Για παράδειγμα, η Βρετανική αμυντική βιομηχανία με την Αμερικανική αμυντική βιομηχανία. Ή μπορούμε να επεκταθούμε ακόμα και, στο Ισραήλ και στην Ινδία. Στις χώρες αυτές δηλαδή που μπορούν να συμβάλλουν στην αμυντική τεχνολογία. Και τέλος κύριε Πρόεδρε, Πρέπει να πω ότι αφού η Γαλλία πλέον έχει μπει πλέον πάλι στην ολοκληρωμένη στρατιωτική δομή του ΝΑΤΟ, η όλη λογική της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας καταραίει. Και νομίζω ότι η πιο αποτελεσματική λύση από οικονομικής πλευράς, και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης που περικόπτονται οι εθνικοί προπολογισμοί στι περισσότερε χώρε του δυτικού κόσμου. Λοιπόν, η πιο οικονομικά αποτελεσματική λύση θα ήταν οι έξι αυτέ χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ να αποφασίσουν να μπουν πάλι στο ΝΑΤΟ, να, να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Η Γαλλία το έχει πράξει αυτό και έχουμε έξι μικρότερα ακόμα κράτη τα οποία δεν ήταν μέλη του ΝΑΤΟ και τα οποία πιστεύω ότι θα πρέπει να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Έχουμε το πρόβλημα της ε, δημοκρατίας της Κύπρου που θα πρέπει να καταλήξει σε μια λογική λύση με την ε, Βόρεια Κύπρο, γιατί σαφώς δεν θα θέλουμε στο ΝΑΤΟ, στους κόλπους του ΝΑΤΟ να βάλουμε και το πρόβλημα αυτό. Πάντως θεωρώ ότι είναι πραγματικά γελίο ότι έχουμε δύο αμυντικούς οργανισμούς αυτή τη στιγμή που απαρτίζονται ουσιαστικά από τα ίδια κράτη-μέλη πάνω κάτω και που δραστηριοποιούν ουσιαστικά στο ίδιο προσκήνιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Λουνατσέκ. Καταρχήν ε, θα ήθελα να πω ότι ο συνάδελφος και ο ε, ε, δεν μπόρεσε να παρευρεθεί γιατί κυρώθηκε η πτήση του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γκάλα για το ότι επισήμανε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει συνέπεια σε όλους τους τομείς της πολιτικής και νομίζω ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο σημείο που θα έπρεπε να είμαστε και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει αυτό το ψήφισμα. Όσον αφορά τα άλλα θέματα τα οποία είναι σημαντικά για μας που θεωρούμε ότι θα πρέπει τα σημεία αυτά να συμπεριληφθούν στο κοινό ψήφισμα για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας. Θεωρώ ότι πρέπει καταρχήν να υπάρξει μια ποιοτική αξιολόγηση της ε, μέχρι τώρα πολιτικής ε, ασφάλειας και άμυνας, γιατί όσον αφορά τους δείκτες επιτυχίας, αναφέρεται εκεί ε, το προσωπικό που αποσπάστηκε, ε, η δομή της επιμελητίας, όμως δεν γίνεται λόγος ε, για την αξιολόγηση αυτής της πολιτικής από το πρίσμα της ασφαλείας, ε, για θετικά και αρνητικά στοιχεία σε σχέση με αυτή την πολιτική. Και αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι κάτι ε, το οποίο μας ενδιαφέρει ως πολιτική άμυνας και ασφάλειας. Και κάτι άλλο να πω, ότι αυτό που ενδιαφέρει τον κύριο Γκαλτιέρη αλλά και πολλούς άλλους εξημών είναι να εξετάσουμε τις επιπτώσεις ε, του ψηφίσματος 1325. Δηλαδή, η σύγχρονη πολιτική ασφάλειας χρειάζεται απαραίτητα και τη διάσταση του φύλου. Κατά τη δική μου άποψη, σε οποιαδήποτε αποστολή ε, θα πρέπει να υπάρχει και ένας σύμβουλος ε, για θέματα φύλου και ε, κάθε εντολή που δίδεται θα πρέπει να περιλαμβάνει και ένα σχέδιο για την υλοποίηση αυτής της εντολής που θα σχετίζεται άμεσα με τη διάσταση του φύλου. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι κατά το παρελθόν αποκλείονται γυναίκες από τέτοιου είδους αποστολές. Ε, πρέπει λοιπόν να συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο γυναίκες και αυτό είναι κάτι ε, που θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας σε σχέση με τις αποστολές. Και κάτι άλλο τι ακριβώς συμβαίνει με το θέμα του αφοπλισμού και με τη μη διάδοση ε, μαζικών όπλων καταστροφής. Ε, τέτοιου είδους ε, θέματα δυστυχώς δεν αναφέρονται. Ας πούμε, η Βρετανική και η Γαλλική πυρηνική γαλλικά και βρετανικά πυρηνικά όπλα. Και εκεί λοιπόν είναι απαραίτητο να υπάρξει αφοπλισμός. Γνωρίζω ότι οι ορισμένοι συνάδελφοι δεν συμφωνούν μαζί μου, αλλά κατά δική μου άποψη αυτό είναι καθοριστική σημασία για να υπάρχει μια ε, κοινή ε, πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Ε, και εδώ λοιπόν, επειδή ετέθη η στρατιωτική συνθήκη, θέλω να πω ότι εμείς επιθυμούμε να ασκηθεί κριτική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτή τη συνθήκη. Γιατί αν θέλουμε και αν έχουμε μια ε, κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας, τότε τέτοιου είδου ε, συμφωνίε ε, θα πρέπει να εντάσσονται στο πλαίσιο τη δομημένη συνεργασίας και όχι σε διμερές επίπεδο. Γιατί είτε θέλουμε αυτή την κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνας, ε, τότε λοιπόν στην περίπτωση αυτή τα ισχυρότερα κράτη-μέλη θα πρέπει να συνάπτουν συμφωνίε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είτε δεν τη θέλουμε αυτή την πολιτική. Ξέρω και η Φανόρντεν ότι εσεί και άλλοι δεν την επιθυμούν αυτή η πολιτική. Υπάρχουν όμω άλλοι, νομίζω η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που επιθυμεί αυτή την πολιτική και γι' αυτό πρέπει να ασκήσουμε τη σχετική κριτική. Τελευταίο θέμα, η ενίσχυση ε, του ε, πολιτικού δυναμικού ε, ως ένα σκέλος των αποστολών. Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα και επειδή αναφέρθηκα και στράφηκα προς τον κύριο Βαν Όρτιν. Η δική του πρόταση για τις έξι μικρότερες χώρες ε, που ε, δεν ανήκουν στο ΝΑΤΟ ε, και εντάσσεται και η δική μου η χώρα, η Αυστρία και λέει ο κύριο Βαν Όρτιν το καλύτερο θα είναι να μπουν οι χώρες αυτές στο ΝΑΤΟ. Κύριε Βαν Όρτιν, αυτό μπορεί να είναι η δική σας η άποψη, αλλά ξέρετε υπάρχει λόγος γιατί αυτές οι έξι χώρες δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Υπάρχει και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια συμφωνία των αδέσμευτων χωρών. ε, το βράδυ ε, έκανα μια συζήτηση πολύ έντονη στην Αυστρία που αφορούσε, είχε ως αντικείμενο την κατάργηση της ε, στρατιωτικής θητείας, αλλά αυτό το θέμα των αδέσμευτων, των ουδέτερων ε, χωρών υφίσταται και οι χώρες αυτές πράγματι θα πρέπει να εντάσσονται περισσότερο στην πολιτική, την κοινή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να στρέφουν την πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερο προ αυτήν την κατεύθυνση, δηλαδή την κατεύθυνση, την πολιτική που ακολουθούν οι ίδιες οι χώρε αυτέ. Μα μένουν 15 λεπτά. σα παρακαλώ λοιπόν να είστε σύντομοι, κύριε Λουζίν. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπορείτε λοιπόν να φανταστείτε, νομίζω, Φαντάζεστε ήδη ότι εμείς ε, όσον αφορά κάποιες ε, διαρθρωτικές προτάσεις για την ε, κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας αλλά και για την ΚΕΠΑ έχουμε άλλες διαφορετικές απόψεις σε επίπεδο αρχής. Ο κύριος Γκαλτιέρη και άλλοι αυτό το θέμα της ασφάλειας το χρησιμοποιούν ως όρο ομπρέλα της ε, πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς όμως έχουμε τελείως διαφορετική προσέγγιση. Εμείς δηλαδή θεωρούμε ότι η εξωτερική, η πολιτική, η εξωτερική πολιτική, η πολιτική ασφάλειας και κυρίως η αναπτυξιακή πολιτική, αυτές οι τρεις ε, πολιτικές ε, πρέπει να παραμένουν ξεχωριστές. Και εμείς επιθυμούμε να επισημάνουμε ότι αν υπάρχει μια τόσο αλληλένδετη εξωτερική πολιτική, τότε δεν είναι δυνατόν να υπάρχει πια αστική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας έχουμε την ε, υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Έχω αναφερθεί επανειλημμένα στο θέμα αυτό. Η διασύνδεση του πολιτικού σκέλους με το στρατιωτικό δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό το θέμα γιατί αυτό σχετίζεται με την υπηρεσία εξωτερικής δράσης αλλά υπάρχουν κάποια δημοκρατικά στοιχεία δημοκρατικής φύσεως, τα οποία δεν εφήγησαν από τους συναδέλφους. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης είναι ένα συγκεντρωτικός μηχανισμός εξουσίας, όπου σχεδόν λείπει. Είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει ο ω ε, έλεγχο. Η Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση ε, σύντομα πρόκειται να καταργηθεί και ω εκ τούτου θα καταργηθεί και η κοινοβουλευτική συνέλευση τη ε, Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση. Σημαντικά στοιχεία τη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση ήδη το 2001 συμπεριλήφθηκαν σε ευρωπαϊκέ δομέ. Στη συνθήκη τη Λισαβόνα αναφέρεται ρητά ότι με τη συνθήκη αυτή δεν προβλέπονται αρμοδιότητε αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου στον τομέα της ε, ΚΕΠΑ και της ε, ε, κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι όσον αφορά την ΚΕΠΑ και την ΕΠΑ, εδώ είχε προγραμματιστεί εκ των προτέρων η κατάργηση του κοινοπτικού ελέγχου, διότι πλέον μιλάμε για διακυβερνητικά στοιχεία της ΚΕΠΑ. Ε, και αυτό που ε, αναφέρθηκε η αλληλένδεση, η διοργανική, αυτή οδηγεί σε έλλειμμα δημοκρατίας. Κυρίως όσον αφορά σε μελλοντικές στρατιωτικές επεμβάσεις, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο δημοκρατικά εκλεγμένο όργανο το οποίο ε, θα μπορούσε να ασκήσει έλεγχο, το οποίο θα μπορούσε να ελέγξει την κατάσταση, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα του, της συναπόφασης. Γι' αυτό λοιπόν εμείς απαιτούμε να υπάρχει κοινοβουλευτικός έλεγχος τόσο της ε, ΕΠΑ, τόσο της ΚΕΠΑ όσο και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Απαιτούμε να υπάρχει πλήρες δικαίωμα ενημέρωσης ε, των κοινοβουλίων των κρατών μελών, δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων, δικαίωμα απόρριψης ε, και ε, μη έγκρισης αποστολών, δικαίωμα ταξιδιού επιτόπου σε περιοχές κρίσης, <clears throat> κάτι το οποίο νομίζω ήδη υπάρχει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξάλλου, ε, τέθησαν και κάποια θέματα χρηματοδότησης. Με τη συνθήκη της Λισαβόνας ε, υπάρχει το περίφημο αυτό Ταμείο Χρηματοδότησης και εδώ θέλω να αναφέρω ότι ο έλεγχος όμως του Ταμείου αυτού δεν αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς λοιπόν είμαστε ρητά κατά της περαιτέρω επέκτασης του κόστους. Ε, και θα ήθελα να φέρω και κάποια άλλα στοιχεία. Ένας τομέας ε, είναι οι ομάδες κρούσης, οι battle groups, ε, κατά πόσον θα υπάρχει μόνιμη δομή συνεργασίας. Το άρθρο 46 εξαιρέθηκε. Είναι το άρθρο αυτό το οποίο αφορά την ασφάλεια εξωτερικής πολιτικής. Κάτι άλλο, ε, ρήτρα ασφαλείας. Και αυτό το θέμα και αυτή η ρήτρα ε, τέθη από ορισμένου συναδέλφους. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι αυτή η ρήτρα ασφαλείας είναι ουσιαστική παρέμβαση στη δημοκρατία των κρατών μελών. Πρέπει να ορίσουμε τι ακριβώς είναι ε, καταστροφή ε, με ανθρώπινη επέμβαση. Με συγχωρείτε πρόεδρε, εγώ έχω το δικαίωμα να μιλήσω όπως και οι άλλοι συντάδελφοι και δεν έχει εξαντληθεί ο χρόνος που προβλέπετε για μένα, γι' αυτό λοιπόν δεν καταλαβαίνω ε, γιατί επιμένετε να συντομεύσω. Εγώ θα πω τις απόψεις μου όπως ακριβώς τις έχω προβλέψει. Κοιτάξτε, υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι που ήρθαν εδώ και θέλουν να καταθέσουν κάποιες, ε, κάποια γενικά σχόλια ε, για την έκθεση του κ. Γκολιατιέρη πρέπει να μας εγκαταλείψει και στις 10.30. Έτσι λοιπόν ε, έχουμε ακόμα 10 συναδέλφους που θέλουν το λόγο. Πολύ ωραία κύριε Πρόεδρε, καλά τα λέτε, αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ, ε, τότε να ε, περιορίζετε τον χρόνο και των προηγούμενων συναντέλφων. Ο Πρόεδρος διαφωνεί και λέει οι προηγούμενοι δεν μίλησαν τόσο πολύ. Θα προσθέσω ορισμένα θέματα, ένα θέμα μόνο λέει ο Πρόεδρος ακόμα, γιατί θέλουν και άλλοι να λάβουν το λόγο. Λοιπόν, θα ήθελα να αναφερθώ ε, σε αυτά που είπε η συνάδελφος Λούνατσεκ και σχετικά με τις αποστολές ε, σχετικά με την ε, βελτίωση του επίπεδου διαβίωση των πολιτών, ε, περαιτέρω εξέλιξη της δημοκρατίας. Θα αναφερθώ και στη διάρκεια και στη συνέχιση όλων αυτών των τομέων έτσι ώστε να υπάρξει ένα στρατιωτικό σύμπλεγμα. Να τονίσω για όλα αυτά. Εμείς είμαστε υπέρ του αφοπλισμού. Εμείς είμαστε υπέρ της μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων. Ο κύριος Μπροκ. Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε ιδιαίτερα ευτυχή θέση γιατί ε, πρέπει να σας πω ότι οι δικές μου θέσεις ε, βρίσκονται κάπου στη μέση ανάμεσα σε αυτά που είπε ο κύριος Βανόρντεν και αυτά που είπε η κυρία Λόζινγκ. Αυτή λοιπόν η θέση της μέσης, του μέσου δρόμου, εμένα πολύ μου αρέσει. Θα ήθελα να συγχαρώ τον συνάδελφο κύριο Γκουαλτιέρη για το σχέδιο που μας παρουσίασε και ίσως ε, μπορεί ένα θέματα να το προβάλλει περισσότερο, αλλά τα βασικά τα έχει παρουσιάσει ήδη. Να σας εξηγήσω λοιπόν γιατί αυτή την ε, κοινή εξωτερική, κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας, γιατί τη χρειαζόμαστε. Τι χρειαζόμαστε διότι εμείς ε, θέλουμε να έχουμε τη δική μας πολιτική ως ήπια δύναμη ο soft power. Ε, αυτό είναι ένα καθαρά ευρωπαϊκό θέμα. Πρέπει να το προβάλλουμε αυτό και να μην ε, εφαρμόζουμε πολιτικέ μόνο μέσα από το ΝΑΤΟ. Μα οι ε, Ηνωμένε Πολιτείε έχουν και δικό του δυναμικό εκτός του ΝΑΤΟ. Όχι μόνο μέσα στο ΝΑΤΟ. Α πούμε, και εμεί θέλουμε στα Βαλκάνια να μπορούμε να διασφαλίζουμε την ειρήνη όταν δεν υπάρχουν εκεί οι Αμερικανοί. Και δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι θα είναι πάντα εκεί οι Αμερικανοί και θα προσφέρονται πάντα ας πούμε, ε, ο γερουσιαστής της Μινεσότα δεν θα μπορεί πάντα να εξηγεί γιατί πρέπει οι δικοί του άνθρωποι να αγγιώνται την ειρήνη στην Ευρώπη. Πρέπει να απεξαρτητοποιηθούμε από αυτό. Και ε, δεν είναι δυνατόν, ε, δεν μπορούμε να αποφύγουμε τις διπλές δομές. Εξάλλου προβλέπεται και στη συνθήκη. Η συνθήκη προβλέπει τη συνεργασία με τον ΝΑΤΟ. Δεν πρόκειται για το Βρετανικό Σύνταγμα είναι κάτι που το προβλέπει η συνεργασία και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Κάτι άλλο που το βρίσκω εξίσου σημαντικό. Χρειαζόμαστε και ένα ευρωπαϊκό, αμυγός ευρωπαϊκό σώμα. Η αδυναμία η δική μας είναι ότι έχουμε ένα σημαντικό εταίρο που ορίζει και εμεί τρέχουμε από πίσω. Χρειαζόμαστε λοιπόν ε, μια... Έχουμε αναπτύξει μια κοινή ευρωπαϊκή ιδέα και στη συνεργασία τώρα που θα έχουμε με τις ΗΠΑ στη νέα αυτή συνεργασία το ΝΑΤΟ ε, θα αποκτήσει μια διαφορετική έννοια και διαφορετικό βάρος. Είμαστε και εμείς η soft power, η ήπια αυτή δύναμη που σας είπα. Και επίσης ε, βλέπω το θέμα το των Γάλλων που μπήκανε στο ΝΑΤΟ, όμως επιθυμούν παράλληλα να αναπτύξουν και την ευρωπαϊκή διάσταση δεν είναι αντιφατικά αυτά τα δύο. Ε, γι' αυτό χαιρετίζουμε την γαλλική πολιτική, την κρίνουμε θετικά. Αγαπητέ κύριε Φανόρντεν, αυτό που είπατε σχετικά με την ε, βιομηχανία άμυνας. Κοιτάξτε, οι επιχειρήσει είναι παντελώς ανεξάρτητες και αυτόνομες. Θα συνεργαστούν με την Ινδία και με όποιον θέλουν. Όμως, αν δεν ε, έχουμε τη δική μας την ευρωπαϊκή προσέγγιση και τα κράτη-μέλη μας είναι ιδιαίτερα αδύναμα, τότε δεν θα υπάρχει πλέον ευρωπαϊκή βιομηχανία άμυνας. Τα εξαρτώμεθα μόνο από τους ε, Αμερικανούς και όποιος εξαρτάται μόνο από τους Αμερικανούς έχει χάσει την πολιτική του ανεξαρτησία. Αυτό λοιπόν πρέπει να το προβάλλουμε. Βεβαίως και πρέπει να ενισχυθεί ο κώδικας συμπεριφορά όσον αφορά την εξαγωγή όπλων. Αυτό είναι μια δυναμία της συνθήκη μας, ότι η εξαγωγή όπλων εξακολουθεί να μην ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει παραμείνει ε, σε εθνική αρμοδιότητα και προφανώς ε, πρέπει όπως σας είπα να υπάρξει ένας καλύτερος ε, κώδικας ε, διοντολογίας. Στον τομέα αυτό δυστυχώς έχουμε αποτύχει. Και τελευταία παρατήρηση κυρία Λούζινγκ. Εγώ δεν επιθυμώ να αποφασίζει η συνέλευση κοινοβουλίων για το κατά πόσον θα επέμβουν στρατιωτικές δυνάμεις ή όχι. Σε αυτή η απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται από κάθε κοινοβούλιο μόνο του. Μόνο του το κοινοβούλιο θα αποφασίζει αν θα στέλνει στρατιωτικές δυνάμεις ή όχι. Εμείς ε, ελέγχουμε ε, τις δαπάνες, αλλά δεν έχουμε τον έλεγχο για το στρατιωτικό στοιχείο, το οποίο αποφασίζεται από, ένα, από κάθε Εθνικό Κοινοβούλιο από μόνο του. Δεν νομίζω λοιπόν ότι μια συνέλευση Εθνικών Κοινοβουλίων μπορεί να αποφασίσει για επέμβαση ε, μάχημων μονάδων ή όχι. Δεν έχουμε ε, φτάσει σε αυτό το σημείο για το πώς κάποιο άλλο θα αποφασίσει αν θα σταλούν οι δικοί μου Γερμανοί στρατιώτε σε ένα ε, σημείο κρίση. Αυτό παραμένει εθνική απόφαση, κυριαρχική απόφαση του ε, κάθε κράτους μέλους. Και εγώ να ενώσω τη φωνή μου με όλους εκείνους οι οποίοι αναφέρθηκαν για, την, για το ενδιαφέρον του κ. Καρτιέρη να παρουσιάσει το θέμα αυτό πριν ακόμα δημιουργηθεί, το, πριν δοθεί το έγγραφο και ότι η ανάλυση η οποία ακούστηκε είναι καθόλου σύμφωνη με τις γενικότερες απόψεις οι οποίες διαμορφώνονται μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας, μετά την προσπάθεια δημιουργίας μιας κοινή ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής είναι λογικό να αναπτύξουμε μια κοινή πολιτική άμυνας ε, σε αυτό το επίπεδο. Συμφωνώ απόλυτα με όσους ανάφερα μια κοινή συμμετοχή όλων των χωρών και αυτό σημαίνει για όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε ανήκουν στο ΝΑΤΟ είτε δεν ανήκουν στο ΝΑΤΟ και παράλληλα θα τόνιζα ότι ορισμένα προβλήματα όπως το προαναφερθέν από τον κύριο Βανόρντεν ε, σε σχέση με την Τουρκία οφείλουν ορισμένες χώρες να συμβάλλουν στην κοινή πολιτική άμυνα και η Τουρκία οφείλει να βοηθήσει στη λύση του κυπριακού προβλήματος, να μην βάζει εμπόδια στην ένταξη της Κύπρου στη PFP, στο Συνεταιρισμό για την Ειρήνη και πολύ περισσότερο να βοηθήσει ούτω ώστε με την αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία να συμβάλλει στο να δημιουργηθεί έναν ενιαίο επίπεδο για την δημιουργία της κοινή πολιτικής άμυνας και ασφάλειας που τόσο σημαντική είναι σήμερα για την Ευρώπη λαμβάνοντας υπόψη και τα γεγονότα στη Βόρεια Αφρική. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, στην αρχή τη συζήτηση, σα είχα πει ότι ο κύριος Γκολτιέρη έχει άλλε υποχρεώσει στι 10.30. Το σημαντικό είναι ότι είχαμε ένα πρώτο γύρο τραπέζι, όλε τι ομάδε που μπόρεσαν να τοποθετηθούν. Στι 28 Φεβρουαρίου θα εξετάσουμε και πάλι την, το σχέδιο έκθεση του κ. Γκολτιέρη. Έτσι λοιπόν σα προτείνω να έρθετε σε επαφή μαζί του για να του κοινοποιήσετε τι θέσει και τι προτάσει σα και θα ήθελα τώρα και ο κύριος Γκουαλτιέρη να πάρει το λόγο πριν να μας εγκαταλείψει και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση στις 28 Φεβρουαρίου αφού θα έχουμε και ένα πρώτο σχεδίο κειμένου. Παρακαλώ. Ρομπέρτο. Συγγνώμη, ένα λεπτό για τον κύριο Βάγκελο από τους φιλελεύθερου γιατί δεν πήρε το λόγο. Ε, ζήτησα το λόγο προηγουμένως, αλλά θα προσπαθήσω να περιοριστώ στο ένα λεπτό αν ε, έχουμε τέτοια κοινή εξωτερική πολιτική όπως έχουμε και σήμερα, δεν χρησιμοποιούμαστε κοινή πολιτική ασφάλειας, ε, γιατί δεν έχουμε καμία κοινή εξωτερική πολιτική. Προς στιγμή συμφωνώ με τον κύριο Πάσκου ότι βρισκόμαστε στο επίκεντρο μιας κρίσης, ε, κρίσης ασφάλειας για την Ευρώπη και μπορεί μόνο έτσι να γίνει αντιληπτή από την Αλβανία φτάνει στον Αγκόρνο Καραμπάχα και στη Δυτική Σαχάρα αλλά και στο νότιο τμήμα. Αν ε, δούμε λοιπόν πώς ε, απαντούν οι πολιτικές ηγέτες, πώς απάντησαν οι πολιτικοί για τις Ευρωπαϊκές Ένωσες τελευταίες μέρες, ήταν η απόλυτη καταστροφή. Όλες ε, οι δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μάλλον ε, έμοιαζαν με σχόλια ανθρωπιστικής οργάνωσης. Θέλω να σας παρατρύνω κύριε Γκολτιέρη να εργαστείτε επί αυτής της σημαντικής έκθεσης αλλά φυσικά συμφωνώ με όλους όσους είπαν ότι έχουμε δύο όψεις του νομίσματος. Ε, αφενός ε, έχουμε τα τεχνικά, οικονομικά ζητήματα και νομικά ζητήματα και έχουμε αφετέρου και το οργανωτικό τμήμα, αλλά έχουμε και ένα άλλο τμήμα που είναι πολιτικό. Και δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία σοβαρή απόπειρα αξιολόγησης ε, των ανοιχτών ε, και κρεμών ζητημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ούτε υπάρχει βούληση σοβαρή συνεισφορά προ την επίλυση των προβλημάτων. Είμαστε σε μια πραγματικά αξιοθρύνητη κατάσταση. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Γκουαλτιέρη. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που πήραν το λόγο. Ζητώ συγγνώμη που πρέπει να καταλήψω τη συνεδρίαση. Απλώ θέλω να διευκρινίσω δύο πράγματα σε σχέση με τα όρια τη έκθεση. Η έκθεση αυτή είναι παράλληλη με την έκθεση Ελμπερτίνη για την εξωτερική πολιτική και την εξωτερική πολιτική ασφάλεια. Έτσι λοιπόν τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ΚΕΠΑ θα συζητηθούν και εκεί. Γι' αυτό και εγώ δεν τα ανέφερα. Τώρα το θέμα που πρέπει να δούμε ε, είναι τι γίνεται με την ε, πολιτική και είναι εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλής μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας και πρέπει να δούμε πώς η συνθήκη της Λισαβόνας μπορεί να αναγνωστεί και κατόπιν πώς μπορεί να συνεισφέρει έτσι ώστε η Ευρώπη να έχει μεγαλύτερες ικανότητες ε, παρέμβασης και μεγαλύτερη ευελιξία στη λογική αυτή της καθολικής προσέγγισης ε, που επιζητά τη χρήση διάφορων μέσων και τη συνοχή τους. Φυσικά, ε, συνοχή μεταξύ των μέσων που έχουν να κάνουν με την πολιτική ανάπτυξη και τις πολιτική άμυνα και ασφαλεία είναι το πρώτο κεφάλαιο και δεν μπορεί παρά να είναι κεντρικό στη δική μου έκθεση. Επίση, θα αναφερθώ στα διμερεί ζητήματα και τη ενισχυμένη συνεργασία. Εγώ φυσικά εύχομαι να αναπτυχθεί η κοινή πολιτική σε μία μόνιμη συνεργασία. Βλέπω ότι σήμερα δεν φαίνεται να υπάρχει στην διάταξη ενεργοποίηση αυτού του μηχανισμού. Και εγώ, ε, αν και αφενός ζητώ την εκπόνηση αυτού του μηχανισμού, υπογραμμίζω και ότι πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένα βήματα. Γιατί αυτή είναι η στιγμή της ανάληψης δράσης. Από αυτή τη σκοπιά διμερείς συμφωνίες μπορούν να είναι χρήσιμες στο βαθμό που ε, μας ε, παρουσιάζουν ότι υπάρχει μια απέτηση και μια δυνατότητα να υπάρχει ε, μια πραγματική συνένωση των μοντέλων άμυνας και κοινή χρήση τους, όμως πρέπει να οδηγηθούμε σε, μια, σε έναν σε μια κοινή χρήση αυτών των μοντέλων. Και σε ό,τι αφορά τα πιο ουσιαστικά πολιτικά ζητήματα, Είδαμε ότι υπήρχε και μια ανταλλαγή απόψεων μεταξύ Λούνατσεκ και Βαν Δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε τα όσα ακούστηκαν. Να πω ότι συμφωνώ με όσο είπε η κυρία Λούνατσεκ σχετικά με την απέτηση να έχουμε μέσα πληροφόρηση που ε, να επιτρέπουν να υπάρχει κοινοβουλευτικό έλεγχο και βάσει τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Έτσι λοιπόν το θέμα τη ενημέρωση ε, θα ε, είναι παρόν στη δική μου έκθεση. Απλώ θέλω να σα πω ότι το Ταμείο Startup προβλέπει ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την ενεργοποίησή του. Έτσι λοιπόν πρόκειται για ένα από τα εργαλεία που, ε, επιτρέπει, το οποίο επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να έχει ένα μεγαλύτερο ρόλο στο στρατιωτικό τομέα. Και ε, πέρα από τη χρησιμότητά του, ε, την πρακτική χρησιμότητά του και γι' αυτό το λόγο πρέπει να ενεργοποιηθεί. Θα στείλω το σχέδιο του κειμένου μόλις ήταν έτοιμο και έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε μία συζήτηση εις βάθος επί του κειμένου. Σας ευχαριστώ. Bien, merci beaucoup. Ευχαριστούμε πολύ. Ζητώ συγγνώμη σε όλους όσους ήθελαν να πάρουν το λόγο και δεν τους τον έδωσα. Πάντως νομίζω ότι τα σημαντικότερα πράγματα υπόθηκαν όσον αφορά την έκθεση αυτή. Στις 28 Φεβρουαρίου θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μια πιο συγκεκριμένη συνάντηση για το ζήτημα αυτό, εφόσον θα έχουμε και το πρώτο κείμενο του κυρίου Γκουαλτιέρη. Ας περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο της μερίσιας διάταξης, με θέμα την έκθεση της κυρίας Κοπά για την μέθοδη πρόσβαση στην κυβερνητική υπηρεσία, η οποία προσφέρεται από το Παγκόσμιο Σύστημα Δορυφορικής Ρεδιοπλοήγησης που προέκυψε από το πρόγραμμα Γκαλιλαίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο μας παρουσίασε το σημαντικότερο τμήμα της πρότασης αυτής. Κυρία Κοπά, έχετε το λόγο για να παρουσιάσετε την γνωμοδότησή σας. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, όπως ε, θυμάστε, τον περασμένο Ιούνιο συζητήσαμε και εγκρίναμε ε, μια γνωμοδότηση σχετικά με την ενδιάμεση αξιολόγηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής πλοήσης, με την οποία καλούσαμε την Επιτροπή ως διαχειρίστρια αυτών των προγραμμάτων να θεσπίσει τους απαραίτητους κανόνες και τις ειδικέ διαδικασίες για την πρόσβαση στην κρατικά ρυθμιζόμενη υπηρεσία του Γαλιλαίου, η οποία είναι γνωστή με το ακρόνιμο PRS, Public Regulated Service. Εφιστούσαμε ιδιαίτερα την προσοχή στην ανάγκη να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, καθώς και να εξασφαλιστεί ένα καθεστώς ελέγχου της μεταφοράς των ευαίσθητων πληροφοριών και της σχετικής τεχνολογίας. Η πρόταση κανονισμού της Επιτροπής, πάνω στην οποία καλούμαστε να γνωμοδοτήσουμε, αφορά ακριβώς την πρόσβαση και τις μεθόδους πρόσβασης σε αυτήν την κυβερνητική υπηρεσία μια υπηρεσία που αποτελεί προστιθέμενη αξία σε σχέση με τις άλλες υπηρεσίες δορυφορικής ραδιοπλοήσης, καθώς πρόκειται για ένα κρυπτογραφημένο σταθερό σήμα προς αποκλειστική χρήση αυτών που ορίζονται ως συμμετέχοντες του PRS. Αυτή στο κείμενο participants, είναι το Συμβούλιο, η Επιτροπή, τα κράτη-μέλη, αλλά και υπό συγκεκριμένε προϋποθέσεις, υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάποια τρίτα κράτη και διεθνείς οργανισμοί. Το ζήτημα φαίνεται τεχνικό. Όμως αυτό το οποίο προσπαθώ με μια σειρά από τροπολογίες που προτείνω είναι να εστιάσουμε σε ορισμένα ζητήματα ασφάλειας που αφορούν στενότερα την υποπιτροπή μας, αλλά και θέτω ένα ζήτημα κεντρικού ελέγχου αυτού του ευρωπαϊκού προγράμματος και επιτήρησης της εφαρμογής των ελάχιστων κανόνων που ορίζονται στο παράρτημα του προτινόμενου κανονισμού. Σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος, με τις τροπολογίες 1 και 10 τονίζω την ανάγκη αποτελεσματικού ελέγχου πρόσβαση στην υπηρεσία και ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των διαβαθμισμένων πληροφοριών του συστήματος. Σε αυτή την υπηρεσία είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχει ανεπιθύμητη πρόσβαση, καθώς και στις ευαίσθητες πληροφορίες του PRS. Με την τροπολογία 2 καταδεικνύω τη σημασία των κρατικών υπηρεσιών του Γαλιλαίου για τις ευρωπαϊκές ε, αποστολές στα πλαίσια της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας και με την τροπολογία 4 τονίζω την ανάγκη έγκαιρης ανάπτυξης δυνατοτήτων για την προστασία των σημαντικότερων υποδομών και κατοχήρωση σταθερότητας και αξιοπιστίας του, συστήμα, του PRS, ειδικά σε περίπτωση διεθνούς κρίσης αλλά όχι Πρέπει να σημειώσω ότι η κοινή δράση 552 του 2004 που αναφέρεται στην πρόταση της Επιτροπής είναι μια σημαντική απόφαση όμως ενεργοποιεί μια διαδικασία για τη λήψη μέτρων αφού έχει προκύψει κάποιο πρόβλημα σε περιόδους διεθνούς κρίσης. Κατά την άποψή μου είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν οι αναγκαίες ικανότητες προτού φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Πέρα από τυχόν επιθέσεις από άλλα κράτη, τρομοκρατικές οργανώσεις, έχει μεγάλη σημασία να εστιάσουμε στους hackers και στους GNSS jammers, που αν δεν ληφθούν έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα μπορούν να πλήξουν την αξιοπιστία ακόμα και αυτού του κρυπτογραφημένου συστήματος. Η τροπολογία 5 υπενθυμίζει τη Γενική Αρχή ότι τα στοιχεία και η τεχνολογία διπλής χρήσης υπόκειται σε έλεγχο εξαγωγών, διευκρινίζοντας έτσι ότι παρά τον αναμφισβήτητα πολιτικό χαρακτήρα του προγράμματος Γαλιλαίο, ιδιαίτερα η τεχνολογία που σχετίζεται με το PRS πρέπει να ελέγχεται και οι εξαγωγές να περιορίζονται μόνο στα εξουσιοδοτημένα τρίτα κράτη. Το άρθρο 2, παράγραφος 7 της πρότασης της Επιτροπής αναφέρει ότι η εξουσιοδότηση αυτή προς τρίτα κράτη ή διεθνείς οργανισμούς προϋποθέτει τη σύναψη διεθνούς συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση η τροπολογία μου αριθμός 9 αποσκοπεί από τη μία πλευρά να διορθώσει ε, κάποιο λάθος του κειμένου τεχνητό και από την άλλη να διευκρινίσει ότι το άρθρο αυτό προϋποθέτει έγκριση εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περνώντας τώρα στο δεύτερο σκέλος της πρότασής μου, θα ήθελα να σημειώσω ότι νομίζω ότι για μας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένα ζήτημα αρχής το Γαλιλαίο είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά συνέπεια είναι σαφές ότι όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα σε όλες τις υπηρεσίες του προγράμματος, εφόσον το επιθυμούν και πληρούν τους ελάχιστους κοινού κανόνες που αφορούν την ασφάλεια και την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το άλλο είναι αυτή η ασφάλεια και αποτελεσματική λειτουργία ε, του συστήματος, ότι είναι σημαντική για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς προβλήματα σε ένα κράτος μπορούν να επηρεάσουν την κατάσταση σε κάποιο άλλο, καθώς βέβαια και να θίξουν την παγκόσμια αξιοπιστία του Γαλιλαίου. Γι' αυτό το λόγο, με τις τροπολογίες μου 3, 11 και 15, τονίζω ότι πρέπει να διασφαλιστεί ένας κεντρικός έλεγχος της εφαρμογής των ελάχιστων κανόνων του κανονισμού και προτείνω έναν πιο ενισχυμένο μηχανισμό επιβολής κυρώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι μόνο σε επίπεδο κρατών μελών δεδομένου ότι αυτός ο οποίος παραβιάζει δεν μπορεί να είναι αυτός ο οποίος επιβάλλει την ποινή. Ιδιαίτερα σε περίπτωση που η μη εφαρμογή επηρεάζει την ασφάλεια σοβαρά του ίδιου του συστήματος η Επιτροπή, σε συνεργασία βέβαια με τα κράτη-μέλη και την εποπτική αρχή του Ευρωπαϊκού GNSS, θα διεξάγουν σε τακτά διαστήματα ελέγχους σχετικά με την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού και των ελάχιστων κανόνων πρόσβασης και ασφάλειας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η Επιτροπή πρέπει να είναι καταρχήν αρμόδια να επιβάλλει κυρώσεις για μη εφαρμογή των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον κανονισμό για τους συμμετέχοντες ενώ τα κράτη-μέλη θα είναι αρμόδια για τον καθορισμό του καθεστώτος των κυρώσεων που επιβάλλονται για τις παραβιάσεις των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται βάσει της παρούσας απόφασης. Με αυτόν τον τρόπο θεωρώ ότι εξασφαλίζεται ένας κεντρικός ευρωπαϊκός έλεγχος, πάντα φυσικά με απόλυτο σεβασμό στην αρχή της επικουρικότητας. Σας ευχαριστώ. Merci Σας ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Ρόιτοβα, που είναι σκιώδη συγητής για το ΕΛΚΑ, μπορείτε να πάρετε τον λόγο στα αγγλικά, γιατί δεν έχουμε διερμηνία στα τσέχικα στην υποεπιτροπή μας. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας πω ότι συμφωνώ με τις περισσότερες τροπολογίες που εξαιρετικά προετοίμασε η συναδελφός μας η κυρία Κοπά. Ωστόσο, έχω κάποια προβλήματα με τα ακόλουθα σημεία. Πρώτον, άρθρο 5 για τις κυρώσεις. Η κυρία Κοπά προτείνει ότι δεν θα είναι τα κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή η οποία θα αποφασίσει ποιες θα είναι οι κυρώσεις οι οποίες θα ισχύουν θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι είδους κυρώσεις μπορεί να επιβάλλει. Γιατί οι ποινικέ κυρώσεις επιβάλλονται σε εθνικό επίπεδο μόνο, είναι εθνική αρμοδιότητα αποκλειστικά. Στη συνέχεια έχω ένα πρόβλημα με την σχετική τροπολογία, γιατί θεωρώ ότι θα προκύψει πρόβλημα σε κοινοτικό επίπεδο όταν θέλουμε να επιβάλλουμε ποινικέ κυρώσει. Δεύτερον, ένα ζήτημα επικουρικότητα που έχει να κάνει με το άρθρο 6, παράγραφος 6, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί εδώ πέρα εξορτημένη πράξη σε σχέση με τα άρθρα 13 και 14, πράξη κάτι εξοδότηση. Και νομίζω ότι εδώ πέρα προβλεπόταν διαδικασία της επιτροπολογίας. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ποιο λόγο προτείνει εδώ τη λύση αυτή, καθότι η διάταξη αυτή, η πρόνοια αυτή είναι προβληματική για το Συμβούλιο. Η ερώτησή μου είναι για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η επιτροπολογία ε, δεν θα ήταν τόσο καλή λύση σε σχέση με τις κατεξοδοτήσει πράξεις που προτείνει πα, παράγραφος 8 τώρα του άρθρου 6. Και εδώ πέρα γίνεται μια αναφορά, πρόβλημα μεταφραστικό μάλλον πρέπει να υπάρχει εδώ πέρα στην τσεχική γλώσσα. Στα αγγλικά πάντως, αναφερόμαστε σε τεχνικούς πόρους της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας, ενώ στα τσεχικά αναφερόμαστε σε τεχνικά μέτρα, technical measures. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω ποια είναι η αρχική πρόθεση της παραγράφου αυτής, της παραγράφου 8. Technical resources ή technical measures, για ποια από τα δύο μιλάμε. Δεν είναι πάντως τόσο σημαντικό το σημείο αυτό. Άρθρο τώρα 8, παράγραφος 5. Ένα πρόβλημα εδώ έχουμε με την εξουσιοδότηση, την αδειοδότηση. Δηλαδή, ένας φορέας ενδεχομένως να χάσει το δικαίωμα αδειοδότησης Επομένως θα πρέπει να διευκρινίσουμε εδώ πέρα ακριβώς ποια είναι η δυνατότητα προσφυγής του φορέα αυτού που έχει χάσει το δικαίωμα αδειοδότησης, που δεν μπορεί πλέον να αδειοδοτηθεί, να εξουσιοδοτηθεί. Ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρθρο 10 τώρα. Και πάλι εδώ πέρα έχουμε ένα πρόβλημα με τις τρίτες χώρες. Και αυτό γιατί νομίζω ότι είναι, είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε πώς ε, μπορούμε να ελέγχουμε καλύτερα το σύστημα. Συμφωνώ με την τροπολογία της κυρίας Σκοπά, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να εμπλακεί περισσότερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην ε, διαδικασία προτιμασίας της συνθήκης για τη λειτουργία, λέω μιλήτρια, συγγνώμη, τροπολογία στην που αναφέρομαι έχει να κάνει με το άρθρο 2 παράγραφο 7. Ξέρω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή και είναι πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορεί να εμπλακεί περισσότερο στη σύναψη συμφωνιών με τρίτες χώρες. Πρέπει όμως να συζητήσουμε και το πώς θα καταφέρουμε να ελέγξουμε καλύτερα τις τρίτες χώρες να υπάρχει και μία επίβλεψη προς αυτές. Και τελευταίο σημείο, στο παράρτημα, παράγραφος 7, Νομίζω ότι εδώ θα μπορούσε να υποβληθεί μια τροπολογία στην οποία θα λέγει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει κάποιες εκθέσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου μας σε θέση να παρακολουθούμε κι εμείς καλύτερα και να ελέγχουμε τη λειτουργία του συστήματος. Ξέρω ότι στο Συμβούλιο υπάρχουν ήδη κάποια προβλήματα όσον αφορά το ζήτημα της επικουρικότητας και κάποια προβλήματα όσον αφορά το ίδιο το παράρτημα. Εδώ πέρα γίνεται μια κοινή αναφορά τόσο στους χρήστες όσο και στις ε, αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση του συστήματος. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι αν θα ήταν καλύτερα να διευκρινίσουμε με έναν καλύτερο τρόπο ποιο είναι το καθεστώς που ισχύει για τους χρήστες και ποιο καθεστώς θα μπορούσε να ισχύει για τις ε, υπεύθυνε αρμόδιες αρχές. Και Σαφώς θα ήθελα να συνεργαστώ με την εισηγήτρια και με τους υπόλοιπους και εισηγητές, κυρία Γκόμες. like thank Να ευχαριστήσω την ε, κυρία Κοπά για, την, ε, πάρα πολύ, για τα πάρα πολύ χρήσιμα στοιχεία που συμπεριλαμβάνει στην ε, πρόταση της Κομισιόν. Πιστεύω ότι επικεντρώθηκε στα πραγματικά ουσιώδη, στη σημασία του Γαλιλαίου για την κοινή μας ασφάλεια και στο εργαλείο PRS και στην αναγκαιότητα να διατηρήσουμε την ακαιρεότητα αυτού του εργαλείου του PRS. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό που αναφέρεστε στην ανάγκη προστασίας ε, κατά των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο που αποτελούν ε, όλο ένα και μεγαλύτερη πραγματικότητα όταν μιλάμε για τέτοια μέσα. Επίσης, νομίζω ότι πολύ σημαντική είναι και η αναφορά στην ανάγκη της διτής χρήσης, των τεχνολογιών ε, διτής χρήσης, και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται ορθά στα εφιστάμενα συστήματα ελέγχου. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και γιατί λόγω ε, οικονομικών ε, περικοπών θα δούμε ότι οι βιομηχανίε μας ε, θα μπουν περισσότερο στον πειρασμό να εξάγουν σε χώρες ε, που μπορεί να αντίκειται στους δικούς μας στόχους με αυτές τις τεχνολογίες. Έτσι λοιπόν, για τις τεχνολογίες της χρήσης ε, προτείνεται η Κομισιόν να είναι αρμόδια για το καθορισμό κυρώσεων έναντι όσων ε, παραμελούν ή στρεβλώνουν το σύστημα PRS. Τώρα για τα σχόλια της κυρίας Ζαϊτόβα. Ναι, φυσικά ποινικέ κυρώσει ε, είναι για τα κρατημέλη, αλλά υπάρχουν και κάποιε κυρώσει που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από την Κομισιόν, οικονομικού χαρακτήρα λόγου χάρη. Ε, επίσης ε, ε, αποκλεισμός από το σύστημα ή αιτήσει για διόρθωση της κατάστασης. Πιστεύω ότι οι προτάσεις αυτές της κυρίας Κοπά είναι ιδιαίτερα ορθές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Λέζινγκ. Ja, vielen Dank. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα να εκφράσω την έκπληξή μου για τη σαφήνεια που περιλαμβάνει η έκθεση της κυρίας Κοπά, αλλά και η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την ε, χρήση του προγράμματος Γκαλιλαίο. Αυτό είναι κάτι που από τότε που είμαι εγώ εδώ στην Επιτροπή ΣΕΝΤΕ, το έφυγα πάντα και η άποψη που εξέφραζα εγώ ότι η στρατιωτική χρήση του Γκαλιλαίου ε, θα μπορούσε να λάβει χώρα. Όλοι μου λέγανε όχι, όχι, όχι, το απέριπταν και τώρα το αναγνωρίζουν ότι 50% του συστήματος Γαλιλαίου ε, θα χρησιμοποιείται για στρατιωτικούς σκοπούς. Και η κυρία Κοπά ε, προέβαλε τη χρήση του προγράμματος Γκαλιλαίου για θέματα ασφαλείας. Αυτό να το επισημάνω λοιπόν ότι βλέπετε από τη μια στιγμή στην άλλη άλλαξε η στάση της Επιτροπής ε, και θα με ενδιαφέρε να μάθουμε πώς έγινε αυτό. Θα με ενδιαφέρε μάλιστα περισσότερο να μου απαντηθεί και το ερώτημα του προϋπολογισμού. Γιατί δεν εξετάζεται ο προϋπολογισμός και γι' αυτό ε, κάνω το εξής ερώτημα. Ένα σύστημα το οποίο κατά πάνω από 50% χρησιμοποιείται για στρατιωτικούς σκοπούς, γιατί να πρέπει αυτό να χρηματοδοτείται από μη στρατιωτικούς προϋπολογισμούς το ότι ε, θα πρέπει να χρηματοδοτεί το πρόγραμμα, αυτό είναι ένα θέμα που Δεν μου έχει απαντηθεί ακόμα η ερώτησή μου. Στην έκθεση της κυρίας Κοπά, το θέμα του κόστους ε, φύγεται πράγματι τον Ιανουάριο. Είχαμε την ενδιάμεση εξέταση του Ευρωπαϊκού ε, Συστήματος Ραδιοπλοήγησης. Είχαμε τη δημοσίευση του συστήματος αυτού και εκεί τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα από ό,τι φοβόμουν. Δηλαδή πλέον στη δημοσίευση αυτή με απόλυτη σαφήνεια αναφέρεται και σας ε, λέω τους αριθμούς ολοκλήρωση του συστήματος 2020 φθινόπορο του 2017 ή του 2018. Επιπρόσθετο κόστος 1,9 δις ευρώ σε ετήσια βάση και στην αρχή θα υπάρξει και επιπρόσθετο κόστος ε, σε τις θέσεις σε λειτουργία. Όλα αυτά τα στοιχεία μπορείτε να διαβάσετε στην έκθεση της Κομισιόν και οι ετήσια τα ετήσια έσοδα ε, μακροπρόθεσμα μπορούν να φτάσουν στα 70 εκατομμύρια. Αυτό αναφέρεται στο θετικό στοιχείο, αλλά για δέστε, συγκρίνω τον αριθμό με το κόστος, μιλάμε εδώ για μια ε, τεράστια επιβάρυνση του φορολογούμενου. Και εδώ να σας πω ότι κάποιος είχε εκφραστεί θετικά για το γερμανικό πρόγραμμα ΟΧΑΜΠΕ. Στην περίπτωση του προγράμματος Γκαλιλαίο ε, είχε αναφερθεί τότε ότι πρόκειται για διασπάθηση του χρήματος του Ευρωπαίου φορολογούμενου. Όλα αυτά που σας είπα τα ήθελα παρακαλώ κυρία Κοπά να τα συμπεριλάβετε στην έκθεσή σας. Ευχαριστούμε. Πρωτού δώσουμε το λόγο στην κυρία Κοπά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριος Στίμαν, παρακαλώ. Yeah, Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που συζητούμε την πρόταση PRS από την πλευρά της Κομισιόν. Ξέρετε, είχαμε μια πρώτη συζήτηση στην Επιτροπή όπου στις 26 Ιανουαρίου εξήγησαμε τη θέση μας. Βασικά είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τις ε, τροπολογίες της Επιτροπής Ήτρε, αλλά και με τις ε, τροπολογίες στην έκθεση της κυρίας Κοπά. Πιστεύω ότι όλα δεύουν προς τη σωστή κατεύθυνση και σκοπεύουν στο να καταστήσουν ε, το σύστημα PRS ε, λειτουργικό. Και ταυτόχρονα αυτό σημαίνει να δίνεται πρόσβαση σε εγκεκριμένου χρήστε, αλλά και να υπάρχει ταυτόχρονα και έλεγχο τη πρόσβαση. Και ε, η Κομισιόν θα βρίσκεται στην καρδιά του συστήματο για να ελέγχει τη χρήση του. Και θα ήθελα τώρα αμέσως να ελθώ στο θέμα που έθιξαν ε, πολλοί αξιότιμοι κύριοι βουλευτές για τις κυρώσεις. Πιστεύω ότι ο όρος αυτός ε, δεν είναι ο καλύτερος πέναλτης. Συνήθως ε, μιλάμε για τη φυλάκιση κάποιου. Δεν είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το ζήτημα αυτό. Έτσι λοιπόν δεν μιλάμε για ποινές υπό το ποινικό δίκαιο νομίζω ότι θα είναι κάτι που θα πρέπει να ρυθμιστεί και εδώ συμφωνώ με την ε, βουλευτή από τη Τσεχία. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να γίνει από τα κράτη-μέλη. Έτσι λοιπόν ε, στην πρότασή μας ε, έχουμε καταγράψει ότι θα πρέπει να ρυθμίζεται αυτό από τα κράτη-μέλη αλλά θα πρέπει να παρακολουθείτε στενά και πρέπει να έχουμε συνεπή λύση. Τώρα, θα αναφερθώ σε αυτά που θα αποκαλούσα εγώ κυρίως διοικητικά μέτρα ε, για να μην υπάρχει πρόσβαση στο σύστημα αν κάποιος ε, το καταχραστεί. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να γίνεται κεντρική διαχείριση αυτής της διαδικασίας, δηλαδή όπως δίνουμε πρόσβαση στους χρήστες θα πρέπει να είμαστε και σε θέση να απαγορεύσουμε την πρόσβαση αν βλέπουμε ότι υπάρχει κατάχρηση. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει ανάγκη αναδιατύπωσης του όρου penalties. Συμφωνώ απόλυτα λοιπόν με τις τροπολογίες όπως σας είπα. Τώρα, για κάποια συγκεκριμένα σημεία που τέθηκαν από τους κύριους βουλευτές. η πράξεις κατανάθεση, κατεξιοδότηση, με συγχωρείτε, ή επιτροπολογία. Το σκεφτήκαμε πάρα πολύ προσεκτικά με τη βοήθεια και της νομικής μας υπηρεσίας αλλά και της νομικής υπηρεσία του Συμβουλίου. Επειδή εδώ μιλάμε για πολύ λεπτομερή τεχνικά μέτρα που θέλουμε να καθορίσουμε, η πράξη κατά εξουσιοδότηση είναι το καλύτερο, με δύο τρόπους. Όταν μιλάμε για τα λέξη στα κοινά πρότυπα, αλλά και στο άρθρο 4, όταν θέλουμε να κοινοποιήσουμε στους χρήστες του συστήματος πώς από τεχνική σκοπιά θα μπορεί να χρησιμοποιείται το σύστημα. Και μιλάμε για πράγματι τεχνικά στοιχεία, για το πώς λειτουργεί στο σύστημα, ποια είναι τα focal points. Έτσι λοιπόν πιστεύουμε ότι η της πράξης είναι το ορθό μέτρο. Σε ό,τι αφορά τώρα στο ESA και την δυνατότητα να υπάρχει κάποια εξουσίδηση του GSA σε αυτό το πλαίσιο πιστεύουμε ότι υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί η τεχνική αρμοδιότητα της GCA της υπηρεσίας. Αλλά και εδώ θέλουμε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί μαζί με το Συμβούλιο Διαπίστευσης Ασφαλείας για να δούμε τι, μπορεί, τι αποτελέσματα μπορεί να έχει το GSA. Επίσης, ε, σε ό,τι αφορά τον έλεγχο ε, εξαγωγών exports control, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο. Για το καθεστώς αυτό, το exports control, Νομίζω ότι έχουμε καταστήσει θέση το πώς μπορεί να αποκλείει ο ένας τον άλλο από το σύστημα. Τώρα για την ε, χρήση τη στρατιωτική του συστήματος. Θέλω να πω ότι ο Γαλιλαίο θα παρουσιάζει πέντε υπηρεσίε. Έχουμε τη μία που είναι η ρυθμισμένη υπηρεσία. Ε, ανοιχτή υπηρεσία, ασφαλεία ζωής, εμπορικές υπηρεσίες, δεν νομίζω λοιπόν ότι είναι σωστό να πούμε ότι το 50% του συστήματος θα χρησιμοποιείται για στρατιωτικούς σκοπούς. Νομίζω δεν ε, αρμόζει να αναφέρουμε το 50%. Και σε ό,τι αφορά τα έσοδα, έχουμε πει στην πρότασή μας, στην πρόταση απόφασης, ότι ο χρήστης θα πρέπει να πληρώνει για το σύστημα. Για η κυβερνητική υπηρεσία, η κρατικά ρυθμιζόμενη υπηρεσία θα πρέπει να χρησιμοποιείται από τις κυβερνητικές υπηρεσίες και για τη διαχείριση καταστροφών και κρίσεων από την αστυνομία και θα υπάρχει τίμημα. Τώρα εδώ δεν είναι το κατάλληλο σημείο να καθορίσουμε το τίμημα. Αυτό θα το αναφέρουμε σε μια άλλη ανακοίνωση όπου θα αναφερόμαστε και στις λοιπές υπηρεσίες και εκεί ε, θα αναφέρουμε και θα καθορίσουμε την πολιτική τιμολόγηση για το σύστημα. Εδώ απλώ αναφερόμαστε στην αρχή ότι ο χρήστη πρέπει να πληρώνει για τη χρήση του συστήματο. Ελπίζω να κάλυψα τα περισσότερα ζητήματα, αλλά ευχαρίστω να απαντήσω και σε άλλες ερωτήσεις αν Ευχαριστώ πολύ για τις διευκρινήσεις. Κυρία Κοπά. Thank you, Mr. President. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους αδέλφους για τη συμβολή τους και προφανώς είμαι στη διάθεσή τους για να συζητήσω μαζί τους και να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε κάποιους συμβιβασμούς. Πρώτον, για την κυρία Μπόιτροβα, θα, Ρόιτοβα, με συγχωρείτε, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε στην παράγραφο 7 του παραρτήματος τροπολογία σύμφωνα με αυτά τα οποία πρότεινε. Είναι πολύ σωστά. Τώρα όσον αφορά τις κυρώσεις. Αυτό το οποίο είχα κατά νου ήταν ένα ζήτημα αρχείας. Θέλουμε μία ευρωπαϊκή προσέγγιση, μία διακυβερνητική προσέγγιση. Πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα ελέγχων. Όπως είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενδεχομένω ο όρος πέναλτης κυρώσεις να αναφέρεται περισσότερο σε ποινικά κολάσιμες πράξεις. Πιστεύω πάντως θα πρέπει να υπάρχει ένα κεντρικό σύστημα ελέγχου για το σύστημα. Θα πρέπει να μπορούμε να έχουμε διοικητικά μέτρα τα οποία θα μπορεί να ελέγχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και να υπάρχει έλεγχο αυτός βέβαια σε περίπτωση παραβίασης. Ενδεχομένως όντως λοιπόν κυρώσεις να ήταν κάπως περιορισμένος. Στην κυρία Λέζινγκ τώρα να απαντήσω. Δεν υπήρξε καμία αλλαγή τοποθέτηση η επιτροπή μα ακόμα όταν και όταν συζήτησε το ζήτημα του Γαλιλαίου πέρυσι. Είχε πει και ψηφίστηκε αυτό και στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια ότι το σύστημα Γαλιλαίο θα πρέπει να υποστηρίζει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και αναφερθήκαμε στην επιχείρηση Αταλάντα η χρησιμοποίηση του Γκαλιλαίου είναι πάρα πολύ σημαντική. Πάρα Επομένως, το Γκαλιλαίο δεν θα είναι ένα σύστημα το οποίο στρατιωτικά θα χρησιμοποιείται για να ενεργοποιηθούν βόμβες, για παράδειγμα. Θα πρέπει όμως, και έχει αποφασιστεί αυτό το πράγμα, να χρησιμοποιείται για να υποστηρίξει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Όσον αφορά τώρα τη χρηματοδότηση του συστήματος, όπως είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο χρήστης είναι αυτός που πληρώνει για το σύστημα και πιο λεπτομερείς διατάξεις ως προς αυτό θα ρυθμιστούν σε ένα μεταγενέστερο στάδιο. Προς το παρόν εμένω στα σημεία αυτά θα έρθω σε επαφή με τους κοιόδης ηγητές προκειμένου να καταλήξουμε σε κάποιους συμβιβασμούς και θα ήθελα και πάλι να σας ευχαριστήσω για τις ιδέες σας και τη συμμετοχή σας. Yeah, merci ναι, ευχαριστούμε πολύ. Η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών είναι 10 Φεβρουαρίου και θα έχουμε δεύτερη ανάγνωση στις 28 Φεβρουαρίου. Σας ευχαριστώ. Αυτά για σήμερα. Έτσι λοιπόν θα συνεδριάσουμε και πάλι στις 28 Φεβρουαρίου. Άννα, να σας ενημερώσω πρόεδρε. Ανησυχώ κάπως γιατί στην Επιτροπή ΛΥΠΕ συζητούμε τώρα μια γνωμοδότηση για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο πρωτόκολλο ε, σε ό,τι αφορά τον έλεγχο της εξαγωγής πυροβολών όπλων για μη στρατιωτική χρήση. Και αυτό το θέμα το συζήτησε εδώ στην, ε, στο Κοινοβούλιο η Επιτροπή Ιντα, γιατί είχε να κάνει με την εμπορία πυροβολών όπλων και τη ΛΥΜΠΕ, των πολιτικών ελευθεριών. Και ανησυχώ μήπω και η δική μα Επιτροπή δεν έχει εμπλακεί. Γιατί δεν έχει εμπλακεί, Γιατί και εμεί έχουμε εδώ εμπειρογνωμοσύνη για το θέμα τη εξαγωγή όπλων. Και ε, φυσικά κάναμε και όλη τη δουλειά που στην κοινή θέση που στο τέλη τη Γαλλική Προεδρία το 2008. Βέβαια εκεί ε, δεν ε, μπορούν να ξέρουν ότι τα περισσότερα πυροβόλα πλά που δεν μπορούν να μην ξέρουν ότι τα περισσότερα που εξάγονται στην Αφρική γιατί αυτά τα όπλα χρησιμοποιούνται σε κάθε είδους ε, σύραξη και χρησιμοποιούνται και από παιδιά και τα λοιπά ξέρετε ότι εξάγονται μέσω της μη στρατιωτικής οδού. Έτσι λοιπόν ανησυχώ Δηλαδή, ουσιαστικά ακολουθείται μια πολιτική διευκόλυνση ε, προκειμένου να προστατεύσουμε τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μας, ενώ κατά τη δική μου άποψη δεν πρέπει να ακολουθούμε αυτή τη γραμμή όταν έχουμε μια καθολική προσέγγιση στα πλαίσια της ε, πολιτικής άμυνας και ασφάλειας. Έτσι λοιπόν ε, θα ήθελα να ζητήσω μήπως να γνωμοποιήσουμε και εμείς για αυτό το πολύ συγκεκριμένο θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα γίνει λοιπόν